Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη. Καθίστε παρακαλώ. Καθίστε γιατί ξεκινάει η ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Sorry being 15 minutes later. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε κατά 15 λεπτά. Ήταν, ξέρετε, η τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών πριν τα Χριστούγεννα. Και θέλαμε να ολοκληρώσουμε όσο πιο πολλά γινόταν. Για όλο το έτος. Τώρα όμως ξεκινάνε οι ψηφοφορίες. Φίλες και φίλοι, σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Πολύ σημαντική ψηφοφορία. Very short. Implementation. Εφαρμογή της πρωτοβουλίας πρίμα σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Προφορική ερώτηση. Συζητάμε. Είναι έτοιμα προφορικής ερώτησης, απάντησης. Συμφωνείτε με την ερώτηση αυτή, όπως προτείνετε. Έναρξη της ψηφοφορίας, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Δεν ολοκληρώθηκε ακόμα η ψηφοφορία. Πέρασε. Τώρα. Πλήρης υποστηρίξη. 48 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Εξαιρετικό αποτέλεσμα, αποδεκτή γίνεται η προφορική ερώτηση λοιπόν. Παρακαλώ, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τις κάρτες σας από το μηχάνημα το συντομότερο δυνατόν τώρα, τώρα. Βγάλετε τις κάρτες σας παρακαλώ. Πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πολύ σημαντικό αυτή τη φορά. Το σημείο 10. Πρόκειται για τον δεύτερο διαρθρωμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαρθρωμένος διάλογος και έχουμε μαζί μας τον κύριο Επίτροπο Κάρλος Μοέδας, ο οποίος ήρθε στην Επιτροπή μας πριν από κάποιες εβδομάδες, στην Ακρόαση, στην πρώτη επίσημη συνάντηση. Τώρα είναι η δεύτερη επίσημη συνάντηση. Τακτική αυτή τη φορά. Με τον Επίτροπο θα έχουμε πολλές στον αριθμό συναντήσεις, ελπίζουμε τουλάχιστον, στην επόμενη θητεία, στην θητεία αυτή. Είσαστε επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία. Πρόκειται για πολύ σημαντικά ζητήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να ανταλλάξουμε λοιπόν απόψεις στο πλαίσιο του διαδρομένου διάλογου με το, μεταξύ Κοινοβουλίου και Επίτροπή για να μα παρουσιάσετε τι προτεραιότητέ σα για του επόμενου μήνε, ιδιαίτερα το 2015. Και θα ήθελα επίση να προσθέσω ότι θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να κατανοήσουμε τι λεπτομέρειε τη έρευνα τη επιστήμης και τη καινοτομία ότι αφορά το νέο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. 315 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ. Και ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε καταρχάς να κοιτάξουμε κάποια χρήματα από το πρόγραμμα Horizon 2020. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε αν τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στον ορίζοντα 2020 ίσως και πιο πολλά χρήματα από ό,τι αφαιρέθηκαν σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση για την ε, κατανομή του κινδύνου. 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ήταν πολύ υποφελής η διαδικασία για τον ορίζοντα 2020 την προηγούμενη φορά. Κάτι παρόμοιο λοιπόν θα θέλαμε να περιμένουμε και αυτή τη φορά. Φυσικά θα έχουμε και άλλα πολλά ερωτήματα. Έχουμε περίπου μία ώρα για τις συζητήσεις μας. Αν ε, μου επιτρέπετε, Επίτροπε, να σας καλωσορίσω εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ε, παρακαλώ να πάρετε το λόγο για μία σύντομη εισαγωγή. Κύριε Πρόεδρε αγαπητέ καθηγητά Μπούζε, αγαπητά μέλη, ε, συνάδελφοι. Χαίρομαι που είμαι και πάλι εδώ σήμερα. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψή μου, όχι ουσιαστικά όμως είναι η δεύτερη, η πρώτη τακτική επίσκεψή μου. Εγώ νιώθω ότι βρίσκομαι εδώ όπως και την πρώτη φορά. Σαν να είναι η πρώτη φορά. Πριν από δύο μήνες, ε, από ό,τι ξέρετε, μου δώσατε πλέον έκτημα την τιμή μου κάνατε να με εγκρίνετε για τη θέση αυτή και είπα ότι ήμουν πρόθυμος να έρθω πολύ συχνά, να έρχομαι πολύ συχνά εδώ πέρα και να κάνω διάλογο μαζί σας. Εδώ είμαι λοιπόν για να συνομιλήσουμε και να σας ενημερώσω για το τι κάνουμε. Όπως ξέρετε ξεκινήσαμε εδώ και ένα μήνα ουσιαστικά τις εργασίες μας, αλλά ήμασταν πολύ δραστηροί και κάναμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι ένα από τα μοτίβα που χαρακτηρίζουν την Επιτροπή σα είναι ότι θέλετε αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να κάνουμε από τις πρώτες εβδομάδες κιόλα. Όπως ξέρετε, υπάρχει στο, Σώμα των Επιτρόπων μια νέα φιλοσοφία πολύ σημαντική για την ετήσια έκθεση ε, ανάπτυξης και για το πρόγραμμα το επενδυτικό στο οποίο θα επανέλθω. Ως επίτροπος που συμμετέχω σε διάφορες ομάδες καθοδήγησης από την ψηφιακή ατζέντα, την ενέργεια, καλύτερη ρύθμιση, γιατί ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περιλαμβάνει διάφορες ομάδες που συνεργάζονται διαρκώς. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να επισκεφτώ τέσσερα κράτη-μέλη, τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία. Και μετέβησα στην Νότιο Αφρική όπου συγκινήθηκα ιδιαίτερα γιατί παρέστησα στην έναρξη του προγράμματος DCPT2 όπου φαίνεται πού πηγαίνουν τα λεφτά των φορολογούμενων για τη διάσωση ζώων πολλών ανθρώπων και με τις πρωτοβουλίες που καταδεικνύουν τις προτεραιότητες του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η πρώτη πρωτοβουλία μου, θα θυμάστε, ήταν ο έμπολα. και το πώς καταφέραμε να πάρουμε 280 εκατομμύρια ευρώ ε, μισά από ιδιωτική και μισά από δημόσια χρηματοδότηση για να γίνουν μελέτες για κλινικές, ε, κλινικά πειράματα και για εμβόλια για τον έμπολα από το ορίζοντας 2020. Και στο κτίριο Μπερλεμούν για να δείξουμε τι γίνεται με το σχετικό scoreboard και να δείξουμε ότι σε ό,τι αφορά θέματα έρευνας και ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά τις δυσκολίες συνεχίζει να επενδύει στον τομέα αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Volkswagen είναι κορυφαία επενδυτρία εταιρεία και είναι από την Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε όμως με το νέο επενδυτικό σχέδιο. Πολύ εξημών είχατε την ευκαιρία να αντιδράσετε στην ανακοίνωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρόεδρο Juncker, από τον αντιπρόεδρο Κατάινεν και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με το νέο λοιπόν αυτό επενδυτικό πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουν μια νέα όθηση στην ανάπτυξη. Το σχέδιο λοιπόν έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου χρειάζεται αυτό ο ενάρτος κύκλο αν θέλετε επενδύσεων αφενό, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική πειθαρχία από την άλλη. Αυτό το τρίγωνο λοιπόν ε, έλειπε. Έλειπε μία γωνία του τριγώνου. Και το σχέδιο το επενδυτικό έρχεται να συμπληρώσει αυτόν τον ε, κύκλο τον ενάρετο που χρειάζεται για να μπει πάλι σε τροχιά ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά παρά το πρόγραμμα επενδύσεων, όλοι νομίζω Ακούσατε διάφορες παρουσιάσεις. Θα ακολουθήσω την πρόταση του καθηγητά Μπούζεκ για να σας ε, παρουσιάσω την οπτική γωνία της έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας. Πώς εμείς λοιπόν τα βλέπουμε όλα αυτά. Αυτό που είχα υπόψη μου για σήμερα είναι να ξεκινήσω απαντώντας κάποιες ερωτήσεις πρωτού καντεθούν, γιατί θεωρώ ότι είναι δίκαιες και θεμητές και με βασανίζουν και εμένα. Να σας δώσω λοιπόν μερικές απαντήσεις και μετά θα κάνετε τις ερωτήσεις σας και έτσι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτό. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που ανέκυψε στο μυαλό μου όταν άκουσα την πρώτη μελέτη του κυρίου Κατάινεν για το επενδυτικό σχέδιο είναι γιατί θα πρέπει ο ορίζοντας 2020 να συνεισφέρει στο επενδυτικό πακέτο. Εδώ ελπίζω να μην χρειάζεται να σας πείσω. Γιατί όλοι κατανοούμε σήμερα στην Ευρώπη ότι ο ρόλο της έρευνας και της επιστήμης και της ε, καινοτομίας είναι πραγματικά κρίσιμος για την ανάπτυξη και για τις θέσεις απασχόλησης. Άρα η συμβολή του ορίζοντα 2020 στο επενδυτικό πακέτο είναι κάτι το υποχρεωτικό. Οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο θα έπρεπε να περιλαμβάνει την έρευνα, την ανάπτυξη, την ε, καινοτομία και την επιστήμη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και νομίζω ότι ως φάκελος, ως χαρτοφυλάκιο και ως μια ιδέα για την Ευρώπη, η έρευνα, η επιστήμη και η κοινοτομία έπρεπε να συμμετάσχουν στο επενδυτικό αυτό πακέτο, μιας και συμπληρώνουν τον ορίζοντα 2020. Δεύτερο ερώτημα το οποίο μου δημιουργήθηκε. Σκέφτηκα, και τι θα γίνει, θα βρεθούμε σε μια θέση όπου ο ορίζοντας 2020 θα είναι σε ανταγωνιστική θέση με το επενδυτικό πρόγραμμα. Εγώ νομίζω ότι είναι σαφές από τις παρουσιάσεις που έγιναν από τον ε, κύριο Κατάινεν είναι ότι η απάντηση είναι αρνητική, όχι, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουν παρομοιούς στόχους μεν. Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, θέσεις απασχόλησης, αλλά ουσιαστικά διαφέρουν, είναι συμπληρωματικά ως προγράμματα. Και αυτό είναι λογικό ότι θα μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο επενδυτικά προγράμματα για να έχουμε καλύτερη, καλύτερα αποτέλεσμα. Αλλά φυσικά νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πραγματικότητα και πάντα θα είμαι ειλικρινής μαζί σας για διάφορα θέματα. Ένα ερώτημα που είναι σημαντικό να διελευκάνουμε αφορά το προφανές. Πώς ο ορίζοντας 2020 μπορεί να συμβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο, ενώ υπάρχουν ε, ελλείμματα στις πληρωμές σε ό,τι αφορά τη λειτουργία προγραμμάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να σας πω τι σκέψεις έχω για το θέμα αυτό. Που είναι ξεκάθαρες πρέπει να ομολογήσω. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση των προβλημάτων αυτών. Είναι ουσιαστικά ε, διτό το πρόβλημα. Καταρχάς, μέχρι το 2014 όπου είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πληρώσει όλου του λογαριασμού που έχει λάβει από τα κράτη-μέλη. Έχουμε συμφωνήσει με τι προθεσμίε και ξέρετε ότι έχει γίνει προσπάθεια από το Γενικό Διευθυντή για να το κάνει αυτό. Γιατί περιορίσαμε την προχρηματοδίτηση, έγιναν κάποιε αναβολέ, προφανώ, αλλά έχει γίνει η δουλειά και έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα για εσά σήμερα. Για το 2015 θα επανέλθω σε αυτά που είπα στην ακρόασή μου. Ότι είμαι αντίθετο σε ό,τι αφορά τις γραμμές για τον προπολογισμό για την έρευνα. Ανεξάρτητα από το ποσό που περιλαμβάνουν. Και μίλησα με την Επιτροπό Τζεοτζίεβα, η οποία είναι πολύ υποστηρικτική και συμφωνεί με τις θέσεις μου. Στην αναθεώρηση λοιπόν για τον προπολογισμό του 2015 θα δείτε ότι έχει διασφαλίσει ότι οι τίτλοι 1α και 1β ε, θα έχουν τους σωστούς πόρους προκειμένου να συνάδουν και με το επενδυτικό πρόγραμμα. Άρα, εδώ χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και όχι μόνο τη δική σας βοήθεια ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σε ό,τι αφορά τη σχέση σας με τις εθνικές σας κυβερνήσεις και με τις πατρίδες σας για να εξηγήσετε τη σημασία όλων αυτών, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη δεν το αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικά είναι τα θέματα αυτά. Και ύστερα έχουμε την ε, ανάθεση των 2,7 δισεκατομμυρίων ε, σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα. Καταρχάς, θα πρέπει να δούμε ότι πρόκειται για ένα τριετές ε, πρόγραμμα έργο πάνω από τρία έτη και τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να καλύψουν ένα δαμείο για τρία, τρίτη περίοδο. Και, και φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει ανάγκη για να γίνει πληρωμές σε, σε χρήματα και δεν θα υπάρξουν ελλείμματα γιατί θα υπάρχει παρατεταμένη χρονική περίοδο. Άρα σε ό,τι αφορά το ρευστό που διατίθεται, θεωρώ ότι είμαστε εντάξει. Τώρα λοιπόν έχουμε το θέμα το εξή. Θα με ρωτήσετε με τη σειρά σας, γιατί δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη απάντηση σήμερα, το πώς μπορούμε να δούμε τον ορίζοντα 2020 και να βρούμε από πού θα βγουν τα χρήματα. Δεν έχω οριστική απάντηση να σας δώσω. Εργαζόμαστε επ' αυτού. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το θέμα αυτό και τι πιστεύετε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα πιθανά σενάρια. Αλλά πάντα να έχουμε υπόψη μας ποιος ήταν ο στόχος των 2,7 δισεκατομμύριων αυτών. Ποιος είναι ο στόχος. Έρευνα. Όχι πιο πολλά επικίνδυνα προγράμματα και μάλλον προγράμματα με ρίσκο στην ανάπτυξη. Ναι. Για την έρευνα και την καινοτομία. Ναι. Τέλος. Και θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα σας αναφέρω στις απαντήσεις μου. Ήθελα να συζητήσω λίγο το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Γιατί θα παραστώ σε αυτό αύριο και ήθελα να σας ε, ενημερώσω για κάποια ζητήματα θα γίνει μια συζήτηση επί της πολιτικής για την επιστήμη, για την κοινωνία και ξέρετε αυτό το θέμα της επιστήμης και της κοινωνίας θα ενταχθεί στην δήλωση της Ρώμης. Θα την υποστηρίξω πλήρης τα συμπεράσματα επίσης ε, του Συμβουλίου για τον χώρο έρευνας που αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας, σας το είπα, η σημασία λοιπόν του οδικού χάρτη για το 2015. Τέλος, θα γίνει έγκριση των συμπερασμάτων των, ε, για την νέα ανάπτυξη και προτεραιότητες για την αύξηση της ποιότητας και τη μεγαλύτερη επένδυση. Στο τέλος θα αναφέρω στο Συμβούλιο ότι ήμουν εδώ όταν ε, ακούσαμε την πλήρη συμφωνία για την πρωτοβουλία πρίμα. Θα έχουμε και τις σχετικές συζητήσεις ε, του Συμβουλίου, τις παρακολουθώ. Θα μου θέσετε όμως το ερώτημα αυτό αργότερα, φαντάζομαι, και δεν χρειάζεται να το απαντήσω. Και τώρα λοιπόν, Πρόεδρε, να προτείνω να δώσουμε το λόγο στους βουλευτές για να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και έχουμε καταρχάς έχουμε τους συντονιστάς και τους αναπληρωτές. Και πρώτος ο κύριος Έλερ για δύο λεπτά, γιατί μου στήσει πάρα πολύ συνάδελφοι το λόγο. Κύριε Έλερ. Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω καταρχάς. Ε, τέσσερις επιτρόπους έχω δει στην πολιτική μου ζωή και κανέναν ε, δεν έχω δει που να ήταν τόσο προετοιμασμένο στι εργασίε του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τόσο δύσκολε συνθήκε. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε για το επενδυτικό σχέδιο. Υπάρχει γενικά υποστήριξη, αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα του γιατί θα πρέπει να βγουν όλα από τον ε, προπολογισμό του ορίζοντα 2020 αυτά τα 3 δισεκατομμύρια γιατί να μεταναμηθούν από τα διευθυντικά ταμεία των ορίζοντα και από το γεωργικό ταμείο. Θα ήταν πιο δίκαιο αυτό, θεωρώ εμάς θα μας απασχολούσε το θέμα του earmarking, της ε, επισήμανσης των κονδυλίων αυτών. Πώς θα διευκρινιστεί ότι στα 350 δισεκατομμύρια θα υπάρξει ίσως τη έμφαση για την έρευνα και την καινοτομία. Ένα τρίτο θέμα είναι το θέμα του προϋπολογισμού. Αν υπολογίσουμε τα 2,7 δισεκατομμύρια, τα 1,1 δισεκατομμύρια περικοπές από το Συμβούλιο, από τα 3,1 που προβλεπόταν για το 2015. Αν δούμε λοιπόν ότι με 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογίες για τα... Α, μας λείπουν 15 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για μείωση τελικά συνολική 25% του ορίζοντα 2020. Να ξέρουν οι συνάδελφοι τι συζητάμε. Διαρκώς σφάζουμε, περικόπουμε Το περικόπτουμε τον προϋπολογισμό για τον ορίζοντα 2020. Αυτή είναι μεγάλη πρόκληση και μια τρίτη ερώτηση. Έχει να κάνει με την ελπίδα μας για την ε, σύνθεση μεταξύ διευθυντικών ταμείων και του ορίζοντα 2020. Πώς συνεργάζεστε με την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο και ποια είναι τα σχέδια προκειμένου να υπάρχει μια συνολική εικόνα για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Ντερούις, από τους Δημοκρατές. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει η κυρία Ρούις. Πρώτα πρώτα το πρόγραμμα, το επενδυτικό του Γιούγκερ είναι θετικά μαντάτα. Και θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, κλίμα εμπιστοσύνη στον δύο τομέα για να έχουμε την συνέργεια δυτικού και δημοσίου τομέα. Πρώτα-πρώτα ε, είπαμε ότι αυτό το οποίο λείπει μια τέταρτη ε, τέταρτη γραμμή του προπολογισμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη. Πάντως, πέραν αυτό, να δούμε το ζήτημα της χρηματοδότησης και πώς όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν το πρόγραμμα για τον ορίζοντα του 2020. Πώς θα έχουμε κάποιο είδους προγράμματα χρηματοδότησης, ακριβώς σαν το πρόγραμμα Juncker. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. το πρόγραμμα Horizon 2020 έχει συγκεκριμένη πρικοδότηση και έχουμε κάποια κονδύλια που θα επιτρέψουν το να υποστηριχθούν κάποια στρατηγικά προγράμματα. Βέβαια θα πρέπει να τροποποιηθεί ο σχετικός κανονισμός. Για να μπορέσουμε να δούμε τι θα αλλάξει από τον πυρήνα του Horizon 2020 στο άρθρο 6 για να καλύψουμε τα προγράμματα που θέλουμε. Αλλά εμείς ανησυχούμε όπως ανησυχεί και η επιστημονική κοινότητα. Να δούμε τι θα γίνει με την χρηματοδότηση κινδύνου. Οπότε θέλουμε να μας καθησυχάσετε τι θα γίνει, θα υπάρχουν αυτά τα ε, συνεργατικά προγράμματα, τι, πώς αυτά θα συνάδουν με το Horizon 2020. Σας ευχαριστώ διακόπτη. Τι θα γίνει με τα προγράμματα που αφορούν τις υποδομές, λέει ο Μιλήτρια, αλλά... Συγχωρείτε, αλλά δυστυχώς πρέπει να σας διακόψω. Ο κύριος Γκρομπάρτσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Εδώ είμαι. Με βλέπετε, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε για αυτή την πρώτη ευκαιρία ε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Ναι, προφανώς οι λεπτομέρειες είναι που είναι δαιμονικές και εκεί βρίσκονται όλες οι δυσκολίες. Ε, πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουν πρικοδοτηθεί σωστά όλα τα προγράμματα. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Ανάπτυξη, οικονομική αύξηση, ανοικοδόμηση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτά είναι βασικές προτεραιότητες, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να ε, γίνουν πραγματικότητα χωρίς δράσεις που τις θεωρητικές αυτές ιδέες να τις κάνουν ε, με φτηνή ενέργεια, με επενδύσεις, με υποδομές, με πόρους που ακόμα δεν έχουν αξιοποιηθεί. Να κάνουν λοιπόν όλες αυτές τις θεωρητικές ιδέες να λάβουν σαρκα και Υπάρχουν κάποιες πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας ας πούμε, που πρέπει να μελετηθεί περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα θέσουμε στους εαυτούς μας, γιατί θέλουμε σταθερούς πόρους. Και πώς θα γίνει αυτό αν δεν υπάρξει διαφοροποίηση. Η αγορά εργασία είναι ήδη, είναι ακόμα μάλλον πολύ εφραστή. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας. Πού θα προωθήσετε σύγχρονες μεθόδους εξόρυξης ε, ενέργειας λόγω χάρη, άντλησης ενέργειας από το σχιστολιθικό αέριο, από τον άνθρακα, από τα πυρηνικά, ποια θα είναι το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στο energy mix, στο ενεργειακό mix. Ε, πρόεδρε, ευχαριστούμε ο κύριος Ντεμπάκερ από την Άλντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σχολιάσω κύριε Επίτροπε λίγο πολύ για τα ίδια θέματα. Νομίζω η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί και ανησύχησαν όταν άκουσαν ότι βάσει του πακέτου Juncker μέρος του Horizon 2020 θα λειτουργήσει ως μόχλευση για να φτάσουμε το 2015 και το 2016 σε αυτά που πρότεινε ο κύριος Juncker. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι απλή. Ξέρουμε ότι όταν θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικέ επενδύσει για να υπάρξει μόχλευση για το, για το πακέτο Juncker, θα πρέπει να υπάρξουν τέτοια προγράμματα που να περιμένει κανεί και απόδοση. Αλλιώ δεν θα υπάρξει καμία επένδυση. Αυτό αντίκειται στη βασική ιδέα του Horizon 2020 για τη στήριξη της βασικής έρευνας που πολλές φορές δεν δίνει καθόλου αποδόσεις οικονομικό κέρδος. Ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω τι είδου προγράμματα εξετάζεται. Και μετά έχουμε χαράξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική αριστεία, ευρωπαϊκή στρατηγική ατομή, όπου νομίζουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει. Εδώ με το πακέτο Juncker τι γίνεται, μια επανεθνικοποίηση αυτών των στρατηγικών, διότι τα κράτη-μέλη θα έχουν τα δικά τους προγράμματα και ξέρω ότι η δική μου η περιφέρεια, η Φλάνδρα, έχει προβλέψει 25 ε, δις προγράμματα. Ε, είναι πολύ δυναμική περιοχή, αλλά φαντάζομαι ότι και άλλες χώρες, Γαλλία ή Γερμανία, θα έχουν ε, τόσο μεγάλη ζήτηση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι μπορείτε για να, να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι η Ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία, η ευρωπαϊκή ε, ανάπτυξη και οι στρατηγικέ του θα επιτρέψουν σε ευρωπαϊκέ εταιρείε να συνεργαστούν με πολυεθνικέ και με τα καλύτερα ερευνητικά Ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη. Ε, on behalf of the Greens, ε, Mr. Από του πράσινου ο κύριο Τούρμε. Ευχαριστώ πολύ. Οι πράσινοι στηρίζουμε την ιδέα του κυρίου Γιούγκερ και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επενδύσει. Όμως για την άρνηση μόχλευσης από το Horizon που σωστά περιέγραψαν ο κ. Έλλερ και ο κ. Κάριν, είναι, είναι ήδη κάτι που μας ανησυχεί και το οποίο είμαστε σύμφωνοι. Δεν ξέρουμε αν από εκεί πρέπει να ε, περιμένουμε στήριξη Πρέπει να πούμε όχι λοιπόν, οι εγγύσει. Πρέπει να πούμε όχι. Υπάρχουν άλλα κονδυλία όπως αυτά των διευθυντικών ταμείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ενεργειακή αποδοτικότητα λόγω χάρη και ως revolving funds ή κάτι τέτοιο αντί να μπερδεύουμε τα πάντα. Νομίζω λοιπόν από κοινού πρέπει να πούμε όχι στην άντληση κονδυλίων από το Horizon 2020 και να δούμε και τα θέματα της ρεσιμότητας. Αυτό που είπε και ο κύριος Ντεμπάκερ, όχι στην επανεθνικοποίηση. Και μια δεύτερη παρατήρηση, το είπα χθε και στον κύριο Κανιέτε, θέλουμε η καινοτομία και η έρευνα να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και τι ευρωπαϊκέ βιομηχανίες. Οι μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις του μέλλοντος θα είναι ανανεώσιμες. Το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Μεταξύ των ανανεωσίμων θα υπάρχει η αιωλική, όπου έχουμε προχωρήσει αρκετά, και η ηλιακή. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την ηλιακή. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο με τα μαχανήματα και του εξοπλισμού, αλλά οι Κινέζοι στο εθνικό του πρόγραμμα λένε ότι 80% του περιεχομένου των μηχανημάτων θα πρέπει να παράγεται σε κινέζικα εργοστάσια και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν προβλέψει 750 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της παραγωγής φωτοβολταϊκών. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να παραμείνουμε πρωταγωνιστές και σε αυτό το θέμα ε, και να συνεργαστούμε κύριε Επίτροπε ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και έρευνα στην Ευρώπη και για τα φωτοβολταϊκά. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε Μουέδας. Είναι μεγάλα τα ζητήματα που τίθενται σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα 2020 και το επενδυτικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ε, λάβουμε μέτρα συγκεκριμένα για να συμφωνήσω με τον κύριο Έιλερ που λέει ότι τα ορίζοντα 2020 ε, θα πρέπει να πάρει ε, κονδυλία και από τα στρατιωτικά προγράμματα και από το Ταμείο Γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι μέτρα θα εφαρμόσετε εδώ πέρα για να μην ε, αδειάσει ο ορίζοντας 2020 για το επενδυτικό πρόγραμμα. Δεύτερο, δεύτερη ομάδα ερωτήσεων. Είναι ανησυχητικό γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια από τα, από τα προγράμματα έρευνας δεν ε, υπάρχουν μάλλον 30, 43% των ε, κρατών μελών πήγαν στη, στα ταμεία αυτά και αυτό το ποσοστό έμεινε, ε, μειώθηκε αργότερα. Ποια μέτρα λοιπόν θα λάβετε ε, προκειμένου τα μέσα να είναι για την έρευνα και την ανάπτυξη πραγματικά και για τις επιχειρήσεις συγκεκριμένα που είναι το 60% του δυναμικού καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, μπορώ να σας ζητήσω να απαντήσετε τις ερωτήσεις. of the political groups. I want to respect the <laughs> um, think... Ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα πρέπει να σας πω ότι ε, είναι πάρα πολύ ευχαριστώ το ότι διαπιστώνω πως όλοι σας προβληματίζεστε και ανησυχείτε για κάποια σημεία τα οποία θεωρώ σημαντικά για όλους μας και πρέπει να τα συζητήσουμε. Και να σας απαντήσω, όχι αν με τη σειρά από πολλές ερωτήσεις, ο κύριος Ντεμπάγκερ είπε ότι γίνεται με τη μόχλευση όσον αφορά τα προγράμματα και νομίζω αυτό είναι μια ωραία ε, αφετηρία για τις ερώτα απαντήσεις. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μένα ως επίτροπο όταν ασχολήθηκα με το πρόγραμμα επενδύσεων ήταν το ότι να εξασφαλίσουμε το πώς αυτό το πρόγραμμα θα σχετίζεται με την ανάπτυξη και άρα αυτό σημαίνει καινοτομία, επιστήμη, παιδεία, έρευνα. Και μια, ένα σημείο, μια διατύπωση στο κείμενο πρέπει να σας πω ότι το, το, ε, έχει λάβει υπόψη ο πρόεδρος κατά και όλοι εάν το διαβάζετε θα διαπιστώσετε ότι ο στόχος ε, του Ταμείου είναι να ε, υποστηρίξουμε προγράμματα σε έρευνα, παιδεία και καινοτομία. Οπότε, το να έχει εντοπίσει ο πρόεδρος Κατάνιεν αυτό το σημείο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείναμε ιδιαίτερα εμείς αυτό και αν θέλουμε να αλλάξει το μοντέλο της ευρωπαϊκής οικονομίας και να δούμε το πώς θα ξεκαθαρίσουμε τα προγράμματα που αποδίδουν αυτά που δεν αποδίδουν, να δούμε πώς θα έχουμε κάποια κριτήρια, κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν όλες τις επενδύσεις, να είναι οι επενδύσεις ε, υποστήριξη των παραγωγικών προγραμμάτων. Αυτό βέβαια ε, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά ελπίζω και διαπιστώνω ότι και εσείς το ίδιο πιστεύετε από όσα είπατε, ότι στις επόμενες φάσεις μετά από το Συμβουλίο θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις κατευθυντήριες για το, για το επενδυτικά ταμείο που θα έχουμε για τους πόρους αυτούς. Οπότε και αυτό θα είναι το εργαλείο για να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα αξιοποιούνται σε προγράμματα για έρευνα, ε, για την ψηφιακή οικονομία, την καινοτομία κλπ. Αυτό είναι το πρώτο, αυτό που θέλω να σας αναφέρω. Και αυτό απαντά σε όσα διατύπωσε ο κύριος Ντεμπάκης. Μετά, είχαμε άλλη μια ερώτηση από τον κύριο Γκρόμπεσιτς. Συγγνώμη που δεν μπορώ να προφέρω σωστά το όνομά σας. Ε, μας μιλήσατε για την ενέργεια και τι θέλουμε να καταφέρουμε σχέση με την ενέργεια και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά την έρευνα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα προκύπτει από τις πρόσφατες αποφάσεις της Ένωσης ότι εστιάζουμε την προσοχή μας σε εκπομπές χαμηλών εκπομπών, διοξιδίου κλπ. Άρα, γι' αυτό έχουμε δεσμευτεί για το ορίζον 2020. Θα πρέπει σε αυτούς τους τομείς να έχουμε την έρευνα ανανεώσιμα, χαμηλές εκπομπές, αποτελεσματικότητα ενεργειακή και αυτά τα είπαμε και όταν είχα την ακρόασή μου ότι είναι σημαντικό, είναι ο ρόλος του δικού μου χρωτοφυλακίου να είμαστε οι φύλακες των ε, επιστημονικών στοιχείων για αυτούς τους τομείς, ας πούμε το σχεσοριστικό αέριο. Ναι, έτσι θα ενημερώνουμε τον κόσμο σε σχέση και με τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι θα είναι η συζήτηση σωστή. Οπότε, έχω δεσμευτεί να επισημαίνω τους κινδύνους που τυχόν αναφύονται. Να ξέρουμε επιστημονικά τι διακυβεύεται. Επίσης, έχαμε την ερώτηση του Κλωτούρμες ρώτησε και το τι κάνουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να, εκεί είναι ο Κλόντ. Με ακούει. Στα γαλλικά θα ήθελα απλώ να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Τούρμες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επαναλαμβάνει ο Επίτροπος. Τονίζοντα ότι πρόκειται οπωσδήποτε για μια προτεραιότητα του προγράμματος Horizon 2020 και σύντομα θα τα πούμε εσείς και εγώ, θα ακούσω και τις δικές σας προτεραιότητες, γιατί αναμφίβολα είναι στα θεματολογία σας πολύ ψηλά, νέοι στόχοι το 2030 για τις ανιώσιμες πηγές και άρα θα πρέπει να εργαστούμε εντατικά στο μέλλον και θα επανέλθω, θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν έχω μαζί μου όλα τα στοιχεία για το τι γίνεται για τις ανανεώσιμες πηγές. Έλες. Έλερ. Μάλλον. Εύστοχο αυτό το οποίο είπατε. Κύριε Έλερ, σας ευχαριστώ. Κατάλαβα καλά. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προβληματισμό μας. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα πάνε σε έρευνα, επιστήμη και καινοτομία αυτά τα χρήματα. Ναι, θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε και ελπίζουμε να βοηθήσει και το Κοινοβούλιο. Ότι δηλαδή στις κατευθυντήριες για αυτά τα χρήματα θα υπάρχει αυτή η δέσμευση. Ότι θα πάνε σε αυτούς τους τομείς. Έρευνα, επιστήμη, καινοτομία. Και το λέω και στον πρόεδρο Κατάνη κάθε μέρα αυτό, όταν το βλέπω. Τώρα είπε και κάτι άλλο ο κύριο Σέλερ. Για το 2-1, 7-1. Τα 2,7 δις αφορούν μια τριετία. δεν υπάρχει κάποια επιπλέον ειδική δέσμευση ότι αυτά θα εκταμιευθούν ε, άμεσα, αλλά τέλος πάντων θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το Συμβούλιο. Επίσης, ο κύριος Σέλερ μας είπε για τα διαπιστωτικά ταμεία και για άλλα κεφάλαια. Ξέρουμε και εγώ και στην Ευρωσκρέτου ότι αυτό είναι κάτι το δύσκολο υπήρχε καθετοποίηση πολύ χρόνο. Και συνεργαζόμαστε για, για αυτούς τους τρεις τομείς, καινοτομία, επιστήμη. Ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και έτσι και θα επανέλθουμε και να σας αποδείξουμε ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. για τα διαρθωτικά. Στα βιολογικά ταμεία έχουμε 100 δι για την επιστήμη, την έρευνα για την κοινοτομία. Αλλά προσπαθούμε τώρα να συναρμόσουμε τις προσπάθειες των συναρμοδίων της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η κυρία Κρέτου και εγώ θέλουμε να προχωρήσουμε και θέλουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις να το καταφέρουμε. Κυρία Καμπεθόν να ρωτήσατε για τη χρηματοδότηση. Είπατε κάποιες ιδέες σημαντικές. Να δούμε τι γίνεται. Με αυτά τα 2,8 δις. Ποια προγράμματα θα καλυφθούν. Και ότι τα κρατημέλη μπορούν να υποβάλουν κάποια προγράμματα που να είναι παραγωγικά να έχουν νόημα για το μέλλον. Θα λάβω υπόψη αυτά τα οποία είπατε, γιατί βοηθάτε τον προβληματισμό μου για να μπορέσω να ασχοληθώ με όλους αυτούς τους τομείς που όπως λέγατε και εσείς αξίζουν, έχουν νόημα. Ξέχασα κάτι. κυρία Κάπολα. Είπαμε για τα διαρθρωτικά ταμεία. Νομίζω τα είπα όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακροσκελέστατος κατάλογος εορτών. Θα έλεγα να τον κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ που συμφωνείτε. Και τώρα 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Η κυρία Ντελκαστή Γιοβέρα. 1,5 λεπτά για να χρόνο. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εσείς δείξατε ότι έχετε τη βούληση και ότι έχετε την επίγνωση για το πρόβλημα το οποίο όλοι σχεδόν βλέπουμε και το, το, το, θίγουμε από την ίδια οπτική γωνία. Τώρα το, αυτό το οποίο θέλω να πω, το είπαν και άλλοι, είναι ότι έχουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση τα οποία βεβαίω και έχουν σχέση με την έρευνα και την καινοτομία. Επομένως ε, αυτή η αφετηρία είναι κάτι που δεν έχει ληφθεί υπόψη, ενώ έχουμε επίγνωση και σε έρευνα και για καινοτομία, όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν. Και να μην έχουμε απλώ κάποια χρήματα τα οποία θα προσθεθούν εκεί πέρα. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία το να ξεκινήσουν με υποστήριξη όλες αυτές τις προσπάθειες. Και κατά κάποιο τρόπο να είναι ε, είναι ξεκάθαρο να είναι αναμφίβολο ότι αυτά τα χρήματα πρόκειται να επιστρέψουν στην ε, έρευνα και κοινοτομία γιατί σε ξαναλέω δεν θέμα ανάκτησης των ε, διατεθέντων πόρων αλλά θα πρέπει να, να διευρυνθεί η ίδια η χρηματοδότηση που προβλέπεται στο ορίζον 2020 και κάπως να καταφέρουμε όσο μπορούμε καλύτερα αυτό με όσο γίνεται πιο λίγα λόγια. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ. Θα τα πω γρήγορα λόγω χρόνου. Επίτροπε, εκτιμούμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεστε στο Κοινοβούλιο με ειλικρίνη εντυμότητα, σαφήνεια και ευθύτητα. Δύο πράγματα. Η σχέση μεταξύ των κονδυλίων της έρευνας και της Ρέτζη θα πρέπει εσείς να δώσετε πολιτικές επιταγές και κατεύθυνση εδώ. Στα κράτη-μέλη οι περιφέρειες πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά και να συμπληρώνουν τα κονδύλια. Ιδάλλως δεν θα τα καταφέρουν. Θα υπάρχει επικάλυψη και άτακτη αντί να υπάρχει συντονισμένη χρήση. Έπειτα για τον προπολογισμό του Horizon 2014-2015. Πρέπει ήδη να σκεφτούμε κάποιες ιδέες για το μέλλον και πρέπει μαζί με το Κοινοβούλιο να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον του Horizon, κύριε Επίτροπε. Και τέλος ένα φιλεγόμενο θέμα. Εκτός είναι σαφέ, σαφές μάλλον πέραν αμφιβολίες ότι έχουν περικοπεί οι πόροι του Horizon και δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, ακόμα και τους ε, ε, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του προγράμματος. Εδώ ας φροντίσουμε τουλάχιστον, εάν πάρουμε 2,7 δις, να γυρίσουν στην έρευνα και την καινοτομία τα διπλά ή τα τριπλά. Να το κάνετε αυτό σε συνδυασμό με τον κύριο Κατάινεν και θα φροντίσουμε και εμείς να το θυμίσουμε σε όλους τους επιτρόπους που θα έρθουν εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σύντομο ομιλία, αλλά πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές. Ο κύριος Χένκελ Αντιπρόεδρος. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι επασκεφθήκατε ήδη τη Γερμανία. Η παρουσίασή σας νομίζω ότι έκανε πολύ θετικές εντυπώσεις για τα θέματα τα οποία ήδη ακούσαμε και από τους άλλους και από τον κύριο Έλλερ. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Δεν έχει νόημα εδώ να τα συζητάμε και να παραπονιόμαστε εμεί στον κύριο και ο κύριο Μουέτα σε εμά σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό για το 2015 και τη μείωση του. Να θυμόμαστε ότι έχουμε και ένα καθήκον στα πλαίσια τη δική μα τη ομάδα να φροντίσουμε όχι μόνο από εμά, αλλά και από τις, ε, τα δραστηριοτικά ταμεία και από το ειρηνικό ταμείο να γίνουν περικοπέ. Ανησυχώ για την διαδικασία follow-up της Μπολόνια που από ό,τι φαίνεται αμφισβητεί τα θέματα εκπαίδευσης ε, των νέων σε ό,τι αφορά την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τα πανεπιστήμια έχουν ήδη τοποθετηθεί. Σας παρακαλώ λοιπόν φροντίστε αυτό το φανταστικό εργαλείο να μην χρειάζεται να θυσιαστεί. Ευχαριστούμε κυρία Κρέλ. Με συγχωρείτε, κάπως πιο καθυστερημένα από ό,τι περιμένατε. Σας ευχαριστώ πολύ και δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω τρεις ερωτήσεις να κάνω. Καταρχάς θα ήθελα ότι το θέμα της ε, έρευνας στον επενδυτικό πρόγραμμα είναι σημαντικό. Αλλά πείτε μου, τι κριτήρια σκοπεύετε να βάλετε στις κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να ξέρουμε το τι, τι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Κατά δεύτερον, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα βασίζεται στη μόχλευση 1 προς 15. Τι αντίληψη έχετε για το θέμα αυτό και πώς μπορεί αυτό στο θέμα της ε, έρευνας να λειτουργήσει. Και σε άλλους τομείς είναι ασαφές, αλλά εδώ μιλάμε για την έρευνα. Για πείτε μου λοιπόν. Είμαι και μέλος της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα συντονισμού στα ταμεία, με τα διευθυντικά ταμεία στα θέματα της έρευνας και με τα υπόλοιπα λειτουργικά προγράμματα. Αυτό επί της αρχής δεν προβλέπεται. Δεν υπάρχει ουσία λοιπόν ιδιαίτερη. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει καλύτερο συντονισμός, καλύτερη σύνδεση από το γενικό κανονισμό προβλέπετε, είναι δυνατόν. Το ρωτάω και το θέτω αυτό το ερώτημα στην Επιτροπή κάθε φορά, αλλά αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα, δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να υπάρχει πιο έντονο συντονισμό. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε κυρία μου, ο κύριο Ζωρίνιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα μιλήσω στη μητρική σας γλώσσα, που είναι και δική μου να χαιρετήσω την ε, επί της αρχής τοποθετησή σας, να μην επιτρέψουμε περικοπές στο Horizon 2020. Μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξή μας. Προφανώς η τελική αξιολόγηση που θα πρέπει να κάνουμε ως προς τους πόρους πρέπει να είναι ποιοτική και όχι ποσοτική. Τα κονδύλια του Horizon 2020, τα οποία είχαν ε, θα χρησιμοποιηθούν ως μόχλευση για το πακέτο Juncker, όπως τουλάχιστον ελπίζετε, είναι κονδύλια τα οποία θα πρέπει να τα συνδυάσουμε με, με σωστούς στόχους, εφόσον χρησιμοποιηθούν στο πακέτο. Τώρα, για αυτό που είπατε κι εσείς και από πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπόθηκε ότι στον τομέα σας υπάρχουν 40.000 εκατομμύρια προθέσεις προγραμμάτων από την Φιλανδία, την Κροατία, την ε, Γαλλία, την Ιρλανδία, την Γερμανία και ό,τι καθεξής από πολλές χώρες. Όμως ε, μόνο η Γαλλία επιτρέπει προβλέπει 24 δις για, τα συστήματα ψηφιοποίησης και ψηφιακής σύνδεσης των σχολείων, εξυγχρονισμού των σχολείων. Τι γνωρίζετε γι' αυτό και πώς βλέπετε αυτήν την δυναμική ζήτηση στον τομέα σας. Ε, ζητώ συγγνώμη, ε, που σε έναν επίτροπο από την Πορτογαλία θα το ένα πορτογαλικό ερώτημα, λέει με Πορτογάλος βουλευτής, πώς βλέπετε το θέμα ότι η Πορτογαλία δεν έχει υποβάλει ακόμη καμία πρόταση. Ευχαριστούμε ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από τρία χρόνια κάλεσα όλες τις καινοτομικές επιχειρήσεις της περιοχής μου και ρώτησα Ποια είναι τα εμπόδια που βλέπετε ότι υπάρχουν, γιατί δεν επενδύεται πιο πολύ στι καινοτομίε. Και αν ακούγατε τι απάντησαν, ήταν πραγματικά επουσιώτη πράγματα. Για παράδειγμα, ένα πρωτότυπο το οποίο παράγεται, δεν μπορεί κανείς να το αφαιρέσει από την ε, φορολογικό του ποσό να το εκπέσει. Η εναρμόνιση λοιπόν στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να περιλαμβάνει την κατάργηση τέτοιων εμπορδίων. Γιατί είδαμε ότι στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες σε διάρκεια σε περίοδους κρίσεως δεν ε, μειώθηκαν οι επενδύσεις, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έρνστ λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ να ξεκινήσω ω εξή. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του κυρίου Γιούγκερ είναι ασταθε. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ποσό, το ξέρουμε όλοι. Αλλά δεν ε, τροφοδοτείται το ποσό αυτό. Και συζητάμε λοιπόν τώρα σήμερα τα θέματα του ορίζοντα 2020 και συζητάμε και τα διευθυντικά ταμεία. Η συζήτηση θα είναι πολύ πιο σκληρή, σας το λέω. Και θα ακούμε πάλι τα ίδια και τα ίδια, ότι είμαστε κατά των περικοπών στα θέματα αυτά. Και δεν θέλουμε να μας αφαιρέσουν κονδύλια. Για τον ορίζοντα λοιπόν 2020 και το επενδυτικό πρόγραμμα μας είπατε ότι είναι συμπληρωματικά προγράμματα. Πείτε μας όμως στην πράξη πώς θα δημορφωθεί τι συζητάμε. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να αναφέρω. Πιστεύω ότι στον τομέα της ε, έρευνας και των επενδύσεων θα πρέπει να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα βήματα. Πολύ μεγαλύτερα βήματα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι το απόλυτο ζήτημα λοιπόν για μας και αν μας ε, παραγωνίσουν ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο δεν θα έχουμε κανένα ρόλο. Νομίζω ότι χρειάζονται πολύ πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις και όχι περικοπές. Ανησυχώ, ανησυχώ ιδιαίτερως. Σας παρακαλώ για τοποθετηθείτε για τα δύο θέματα αυτά. Thank you very much, madam, for your... Σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Κάριντς. Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μία ερώτηση που τέθηκε και προηγουμένως και ήθελα να την ε, συνδυάσω με τη δική μου. Θα προσπαθήσω να το πλουστεύσω γιατί το ε, έθεσαν πολλοί συνάδελφοι με διαφορετικούς τρόπους. Δεν κατάλαβα να απαντήσατε, αλλά θέλω να το καταλάβω. Το πακέτο Juncker ζητά πολύ έντονες και μεγάλες επενδύσεις στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει χρήση κάποιων κονδυλίων ε, από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας. Ίσως και να δουλέψει αυτό. Όμως ε, κάποια κονδυλία θα έρθουν από το πρόγραμμα 2020 που όπως δηλώθηκε πολλά από αυτά είναι για τη βασική έρευνα. Ξέρουμε όμως ταυτόχρονα ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να έχουν και δυνατότητα κερδοφορίας. Ιδάλλως γιατί ένας ιδιωτικός επενδυτής, ε, μια οποιαδήποτε εταιρεία να επενδύσει σε κάτι που δεν θα δώσει οικονομική, οικονομικό κέρδος. Ποια είναι λοιπόν τα δύο σενάρια ή μήπως υπάρχει και ένα τρίτο. Τέτοιες επενδύσεις δεν θα γίνουν ή οι επενδύσεις θα γίνουν και θα είναι και κερδοφόρες αλλά δεν θα γίνει έρευνα έρευνα. Τι από όλα αυτά ισχύει. Νομίζω ότι αν το γράφατε θα ήταν πιο απλό. Αυτά από τη σκοπιά των ερωτήσεων για σήμερα. Αγαπητοί βουλευτέ, σα ευχαριστώ για τι ε, ερωτήσει σα και επιτρέψτε μου να αρχίσω στα πορτογαλικά. Γιατί στα πορτογαλικά με ερώτησε ο συμπατριώτη. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω, όπως είπατε και στην παρέμβασή σας, είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε στόχους και να δούμε τι output, τι αποτέλεσμα περιμένουμε από τα διάφορα προγράμματα. Όντω έχουμε, έχουμε λάβει καταλόγους από τις διάφορες χώρες, αλλά πρέπει να αναλυθούν, θα τις φιλτράρουμε τους καταλόγους αυτούς για να δούμε τι προγράμματα έχει νόημα να στηρίξουμε, για να δούμε τι είναι και παραγωγική έρευνα μέσα από όλα αυτά θα πρέπει να δούμε αυτούς τους καταλόγους ως καταλόγους προθέσεων ε, που έχουν καταρτιστεί από τις χώρες. Αλλά θα είναι πάρα πολύ δουλειά για να ορίσουμε στόχους κατευθυντήρες γραμμές ώστε τελικά να παραμείνουν ε, τα πρόγραμματα αυτά. Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτούς τους καταλόγους ε, στην αξία όψεως που μπορεί να έχουν όπως λέμε στα πορτογαλικά και στα αγγλικά. Είναι πάντως ιδιαίτερα σημαντικό τα ίδια τα κάτι μελη και εδώ οι ευρωβουλευτές έχουν ρόλο να διαδραματίσουν. Θα πρέπει λοιπόν τα κάτι μελη να την πολιτική σημασία αποστολής προγραμμάτων, προγραμμάτων για την τεχνολογική γνώση, για την παραγωγικότητα των ίδιων των χωρών. Διότι εάν τα ίδια προγράμματα ε, που έχουν ήδη εκτελεστεί στο παρελθόν δεν θα έχει αυτόν τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στο κέρδος το όλο πακέτο. Στα αγγλικά εκκρεμεί ένα άλλο ερώτημα το οποίο αφορά διάφορους βουλευτές. Κυρία Κρέλ το ανέφερε, μας είπε για το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, ο κύριος Κάρινς επίσης το έφεξε κάπως αλλιώς και απλώς θα ήθελα να σας ε, απαντήσω ε, επί τη βάση της λογικής της αποτελεσματικότητα τη αγορά. Γιατί όταν μιλούμε για πολλαπλασιαστή 15, δεν αναφερόμαστε μόνο σε ένα αριθμητικό στοιχείο, αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικά. Ε, αν έχουμε προαπλασιαστεί τρία για όλα όσα έχουν σχέση με δάνεια και χρηματοδότηση και προαπλασιαστεί πέντε που θα αφορούσε τον ιδιωτικό τομέα και άλλους πόρους, άλλα κεφάλαια τα οποία θα ενεπλέκονται. Άρα δεν είναι λοιπόν ένα μεγάλο νούμερο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Φανταστείτε ένα έργο, ένα πρόγραμμα που βάζει κανείς από τον δημόσιο κορβανά ένα ευρώ και αυτό όμως ενδιαφέρει και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, εάν η αγορά εξετάζει τα προγράμματα στους τρεις τομείς που είπαμε, έρευνα, ε, καινοτομία κλπ, τότε θα πει ότι ένα έβαλε εσύ κράτο, ο ιδιωτικό τομέα θα πει βάζω κι εγώ άλλα 5 ευρώ. Οπότε μπορούμε έτσι να αμοχλέψουμε αυτές, αυτή τη δυτή χρηματοδότηση και να χρησιμοποιήσουμε τον πολλαπλασιαστή 3. Και οπότε πάμε 3 επί 5, 15. Τόσο δεν είναι. Άρα είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί αυτό. Είναι τεχνοκρατικό το θέμα, αλλά όταν μιλάμε για συντελεστή ή πορεπλασιαστή 15, ε, αφορά αυτό ένα χρέος, μια οφειλή, ένα δάνειο, αλλά ο πολλαπλασιαστής είναι μείγμα ιδιωτικής επένδυσης και πόρων. Επομένω, πολύ σωστά όλα αυτά, γιατί ε, όσον αφορά τη διευκόλυνση κατά του κινδύνου, έχουμε ένα δις ε, από την Ένωση, ένα δις από την Τράπεζα Επενδύσεων και μπορεί κανείς να πάει μέχρι τα 15. Έχουμε βέβαια το πακέτο για την καινοτομία και εκεί έχουμε 8 δις, τα οποία είναι από τον δημόσιο κορμανά και άλλα 4 ε, από τα κράτη-μέλη, τώρα σας τα λέω αυτά από μνήμες. Οπότε πάμε το περίπου στα 22. Ε, οπότε όλα αυτά έχουν μοχλευθεί ως ιδιωτική επένδυση. Συγγνώμη αν σας τα λέω πολύ τεχνοκρατικά, αλλά είναι απαραίτητο να σας τα αναφέρω έτσι. Πάντοτε είναι αντικείμενο επικρίσεων ε, ο παροπλασιαστής, αλλά τι να σας πω την του. Κύριε Κάριν, τι θέλετε. Ναι, πέστε μας πιο συγκεκριμένα. Ναι, όλα όπως μας είπατε είναι υπέροχα λογικά. Η ερώτησή μου είναι γιατί έχουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο που αφορά, ε, αφορά ένα πρόγραμμα που δεν θα έχει απόδοση. Γιατί να το κάνει αυτό ο ιδιωτικό τομέα, γιατί να επενδύσει κάπου που δεν θα κερδίσει τίποτα, γιατί να υπάρξει τέτοιου είδου κεφάλαιο. Συγγνώμη, συγγνώμη πρόεδρε, η πρώτη μου φορά είναι, τα χαμένα. ανοιχτή συζήτηση. Όποιο θέλει ό,τι θέλει στον Επιτρόπο. Συγγνώμη, συγγνώμη πρόεδρε. Είδα ότι ε, ο κύριος Κάριν ε, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο όταν τα αυτά. Τέλος πάντων, με αυτό που με ρωτάτε, μπορώ να προχωρήσω λίγο παραπάνω στην επιχειρηματολογία. Ότι δηλαδή ο ιδιωτικό τομέας, εάν θέλουμε να συμμετάσχει στις επενδύσει, τότε η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να στηρίζεστε σε τέτοιου είδους προγράμματα. Φυσικά δεν είναι ανόητοι του ιδιωτικού τομέα να πάνε κάπου που έχουν χαμηλότερη απόδοση. Γι' αυτό νομίζω ότι μας βοηθά για έρευνα και καινοτομία και επιστήμη να το ιδιωτικό τομέα για εδώ και όχι αλλού, γιατί αλλού δεν θα πάει ο ιδιωτικός τομέας. Ναι. Το μήνυμα αυτό το οποίο είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Τόια. Είπατε τι γίνεται με τους πόρους για την έρευνα, τι γίνεται με το διορθωτικά ταμεία και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε. Δίκιο έχετε. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και επίσης του πώς θα έχουμε κίνητρα από τη βάση προς την κορυφή. Παντού. Αυτά λέμε και στην υπηρεσία μου και στην υπηρεσία της κυρίας Κρέτου και προσπαθούμε όλα αυτά να τα διατυπώσουμε και εγγράφως και τελικά όλα αυτά να τα υλοποιήσουμε. Άρα, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και σύντομα θα έρθω στο κοινοβούλιο πάλι και να σας πω πώς ακριβώς θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Άλλη ερώτηση, τον κύριο Μπολόνιο. θα επανέλθω για να σας απαντήσω γιατί τώρα δεν έχω αυτά τα στοιχεία. Όπως ξέρετε είναι κάτι διακυβερνητικής υφής και φύσεως. Δεν είναι θέμα μόνο των 28, αλλά υπάρχει συμβολή της Ένωσης και σίγουρα βοηθά. Αλλά πάντων δεν μπορώ να σας πω κάτι ακριβέστερα, γι' αυτό και θα επανέλθω και θα σας πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις τώρα από τον κύριο Μάνκα, την κυρία Έρνστ, σε σχέση με το με τις επενδύσεις ότι το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες οι χώρες να άρουν τους φραγμούς που εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπορεί κανείς να προτίθεται να επενδύσει άπειρα λεφτά στην επιστήμη και στην έρευνα, αλλά οι χώρες θα πρέπει να έχουν την ευελιξία ε, να προχωρήσουν και να άρουν αυτούς τους φραγμούς. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις. Οπότε αυτό έρχεται να συμπληρώσει, να απαντήσει σε αυτό το οποίο θέσατε. Αυτά είχα να σας πω. Αν κάτι παρέλειψα, σημαντικό, παρακαλώ στείλτε μου ένα email ή αν ξέχασα κάτι θα το συμπληρώσω. Πρόεδρος. Από ό,τι βλέπω όλοι είναι ικανοποιημένοι, λέει ο Πρόεδρος. Α, και κάτι άλλο για την κυρία Καστήλιο. Είπατε ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, να επενδύσουμε. Και με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα να ενισχύσουμε το ορίζοντα 2020, όχι να το αποδυναμώσουμε. Σίγουρα. Και Εγώ αυτό θέλω να γίνει και αυτό και θα κάνω. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτροπέ. Ήταν ε, η πρώτη βαθιά ανταλλαγή απόψεων. Βέβαια, βαθιέ ανταλλαγέ απόψεων είχαμε και στις ακροάσεις. Τώρα έχουμε μια δεύτερη συνάντηση μαζί σας. Συγχαρητήρια για τι απαντήσει σα. ευχαριστούμε πολύ. Uh, Συνάδελφοι, να πω το εξής. Επόμενο σημείο στην εμεί διάταξη Επόμενο σημείο 11. Δημιουργία και λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2037 του κυρίου Ταγιάννη. Αυτό θα το δούμε στις 4 το απόγευμα. Στην απόγευματινή μας συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 3 με ευκαιρίε πράσινη ανάπτυξη για τις ΜΜΕ. Συνάδελφοι, μισό λεπτό, ένα λεφτάκι. Ξεκινάμε στις τρεις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ε, μικρομεσαίες. Τέσσερις. Έκθεση Ταγιάννη. Και στις πέντε Παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα Δόκτωρα Ορμπάν Ρουσνάκ, σχεδιασμός για το Διεθνή Χαρτί Ενέργειας 2015. Αυτά είναι τα θέματα μας για σήμερα. Και τώρα έχουμε ένα τεράστιο διάλειμμα για φαγητό. Σας ευχαριστώ. Um,